Να σας ενημερώσω ότι η επόμενη συνάντηση θα γίνει αύριο, 3 Φεβρουαρίου, στις 9 με το 10.30 και μετά από τις 3 έως τις 11 το βράδυ. Αύριο λοιπόν Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου. Η ημερήσια διάταξη έχει ήδη δημοσιευθεί, βρίσκεται και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό λοιπόν είναι το τέλος της σημερινής συζήτησης. Καλό βράδυ.